σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε να κάνουμε με τις σύντομες παρουσιάσεις ε, των ακολούθων εκθέσεων. Έκθεση της κυρίας Κούνεβα σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ε, σαν οικιακές βοηθοί. Έχετε το λόγο κυρία Κούνεβα. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οικιακό προσωπικό και προσωπικό φροντίδας. Τους επιστευόμαστε τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους αρρώστους μας. Μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την καριέρα μας και να απολαμβάνουμε την κοινωνική ζωή μας, αλλά είναι αόρατοι, αντίλωτοι, ανασφάλιστοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι. Και είναι κυρίως γυναίκες. 2,5 εκατομμύρια οικιακά εργαζόμενοι στην Ευρώπη εκ των οποίων 88% είναι γυναίκες. Δουλεύουν ατέλειωτες ώρες, χωρίς άδειες, χωρίς ετροφαρμακευτική κάλυψη, χωρίς συντάξεις. Δουλεύουν σε συνθήκες που δεν μπορούν να ελεγχθούν γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλοι μέθοδοι επιτεωρήσεις για να τις εντοπίσουν και να τις προστατεύσουν όπου χρειάζεται. Ο πληθυσμός μας που γερνάει και η είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασία δημιουργούν μεγαλύτερες ανάγκε οικιακό προσωπικό και προσωπικό φροντίδα. Τα κράτη-μέλη το γνωρίζουν, αλλά επιτρέπουν να καλύπτονται τα κενά στο πλαίσιο της παραοικονομία. Μειώνουν τις δημόσιε δαπάνε και εκμεταλλεύονται τα κύματα μεταναστών ω νέο φτηνό εργατικό δυναμικό που καλύπτει τέτοιε ελλείψεις. Χρειάζεται άμεσα καταγραφή της κατάστασης στα κράτη-μέλη, επαρκής νομοθεσία για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για αποσχολούμενους σε οικιακές εργασίες που αντιμετωπίζει τις ανάγκε τους συνολικά επαγγελματοποίηση και πιστοποίηση. Η οθέτηση των καλών πρακτικών, η Γαλλία και το Βέλγιο αποτελούν παράδειγματα με διαφορετικό τρόπο. Προσέγγιση από τα συνδικάτα, γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν που να προσφύγουν. Έλεγχη με σεβασμό της ιδιωτικότητας. Ενημέρωση των εργαζομένων τα δικαιώματά τους και των εργοδοτών για τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την συνεργασία που είχαμε την Τάνια Γκονζάλες που συνέταξε την νομοδότηση για την Επιτροπή Απασχόλησης και Οικονομικών Υποθέσεων και όλους τους φορείς που συμβάλλαν στην ανάδειξη του θέματος. Χρειαζόμαστε τη στήριξή τους, ιδιαίτερα τώρα, πριν την ψηφορία της έκθεσης αύριο γιατί η συντηρητική πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ζητήσει ξεχωριστή ψηφοφορία για πολλά και σημαντικά σημεία της έκθεσης, ώστε καταψηφίζοντάς τα να την αποδυναμώσουν. Αν η συντηρητική πλειοψηφία δεν θέλει κανένα δεσμευτικό μέτρο, αν δεν θέλει να γνωριστεί το επάγγελμα, αν δεν θέλει να έχουν δικαιώμα οι εργαζόμενοι ώστε σε συγκεκριμένο χρόνο εργασία, ούτε σε ιατρική κάλυψη, ούτε σε άδεια μητρότητα, αν δεν θέλουν να επικυρωθεί η σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τότε να παραδεχτούν πως θέλουν αντίλωτους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Να πούν ξεκάθαρα πως οδηγούν στη διάκριση των πολιτών σε προνομιούχους και δεύτερης κατηγορίας, πως δεν τους ενοχλεί η εκμετάλλευση των μεταναστριών. Η Ευρώπη καταραίει κοινωνικά και αυτό απομακρύνεται από τους πολίτες της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μερίδιο ευθύνες γι' αυτό. Το ζήτημα που συζητάμε αποτελεί πρώτιστος θέμα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ο Αντών Τσέχοφ έγραψε στον αδελφό του. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι πρέπει κατά τη γνώμη μου να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια. Να σέβονται τα ανθρώπινα όντα ως άτομα. Και είναι η προσωπική ευκαιρία του κατένος και κάθε μίας από εμά να αποδείξουμε ποιος είναι ο πολιτισμός μας και ο σεβασμός μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Τόμκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την εισηγήτρια μας, την κυρία Κούνεβα. Οι στατιστικές δείχνουν μια πολύ δυσάρεστη εικόνα πολλοί και κυρίως γυναίκες εργάζονται ως οικιακοί βοηθή. Δεν είναι όμως μόνο μετανάστες που εργάζονται ως οικιακές βοηθή. Ε, υπάρχουν γυναίκες που ενώ είχαν δουλειά την εγκατέλειψαν για να φροντίσουν την οικογένειά τους, τους ηλικιωμένους γονείς τους, ε, να αναθρέψουν τα παιδιά τους, γιατί δεν έχουν άλλη δυνατότητα. Ε, γιατί η βρεφονιπιακή σταθμοί κοστίζουν. Οι, η ευγυρία ε, είναι πλήρε. Και μάλιστα αυτέ οι γυναίκε, ενώ δουλεύουν στο σπίτι, ούτε κάνουν να γνωρίζει τη δουλειά του, ούτε αμείβονται για αυτήν, ούτε τη χάνουν κάποια κοινωνική προστασία ή ασφάλιση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κάποιε χώρε μέλη και η δική μου, η Σλοβενία, έχουν κάποια μέτρα, έχουμε έναν κανονισμό που διέπει αυτά τα θέματα, αλλά χρειαζόμαστε κάποιε συστημικέ λύσει. Νομίζω ότι πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε με συστημικές λύσεις. Να μειώσουμε την παραοικονομία, κάτι που θα ωφελήσει όχι μόνο τις άνδρες και τις γυναίκες, αλλά το σύνολο της κοινωνίας. Thank you very much and thank you. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και την εισηγήτριά μας για την έκθεσή της και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που υιοθέτησαν πολύ προοδευτικές και συμπονετικές απόψεις. Είναι σημαντικό να διατρανώσουμε στη συζήτηση ότι η κατάσταση των γυναικών που παρέχουν φροντίδα επηρεάζεται από τις επιζήμιες πολιτικές λιτότητας, από την περικοπή των κοινοφελών υπηρεσιών και των δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και στην συντηρητική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και όταν αναγκάζονται οι γυναίκες ε, να παράσχουν φροντίδα στην οικογένεια, αλλά δεν αναγνωρίζονται ούτε υποστηρίζεται, ε, γινόμαστε μάρτυρες μιας παλινδρόμησης ε, και μιας ε, αρνητικής μεταχείρισης ε, των γυναικών. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές. Ούτε καν η ψυχολογική τους υγεία δεν λαμβάνεται υπόψη στην έκθεση. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών για να τηρηθούν ότι παρέχοντας φροντίδα ε, και να αναγνωριστούν. Επίσης, να ε, ενισχύσουμε τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά για να δράσουν και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους χρήζοντες ανάγκη και τα πιο ευάλωτα άτομα. κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, αφού ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κούνεβα, για την έκθεσή της, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με επισφαλείς συνθήκες εργασίας δεδομένου ότι οι οικιακές εργασίες εκτελούνται με τη μορφή της αδήλωτης εργασίας και δεν καλύπτονται από την εργατική νομοθεσία. επιπλέον συχνά δεν υπάρχει κοινωνική προστασία και κάλυψη για τα εργασιακά τους δικαιώματα με αποτέλεσμα οι μισθοί των γυναικών στους τομείς αυτούς να είναι χαμηλοί και να μην τους εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής ειδικά σε χώρες όπως η ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια λαμβάνοντα υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών εργαζομένων που καταπατώνται από την οικονομική κρίση και την έλλειψη νομοθεσία σε ορισμένα επαγγέλματα θα πρέπει οι χώρε τη ευρωπαϊκή ένωση να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των γυναικών που απασχολούνται στι οικιακέ εργασίε και να τι συμπεριλάβουν στην εθνική του νομοθεσία. παράλληλα θα πρέπει να σταματήσει η ευρωπαϊκή ένωση να φτωχοποιεί τι χώρε του νότου και να πλήττει έτσι τα δικαιώματα των γυναικών τόσο σε εργασιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια πρώτα, την κυρία Κούνεβα, για την έκθεσή της για τους οικιακούς βοηθούς και παρέχοντας φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ κατέθεσα 17 δικές μου τροπολογίες στη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Απασχόλης και χαίρομαι ιδιαίτερως που ε, σχεδόν όλες οι ιδέες μου περιληφθήκαν στην τελική μορφή της έκθεσης. Κυρίως ε, η έκκληση να, εγκριθεί, να ε, κυρωθεί από τα κράτη-μέλη η σύμβαση της ΔΟΕ υπερθμών 189 για τις κακούς βοηθούς. Και μάλιστα η Ιρλανδία ήδη έχει κυρώσει τη σύμβαση του ΔΟΕ, αλλά 22 άλλες χώρες μέλη δεν έχουν ακόμη προβεί στην κύρωση και θα πρέπει να το κάνουν επιγόντως. Χαίρομαι που η ιδέα μου για την εξασφάλιση της επαγγελματοποίησης ε, του τομέα αυτού και προκειμένου να ενισχυθούν οι αξιοπρεπείς θέσεις επασχόλησης επίσης περιλήφθηκε στην τελική έκθεση. Και μάλιστα και η έκκλησή μου για να σταχθεί μια οδηγία για τους παρέχοντες φροντίδα και τους οικιακούς βοηθούς στην έκθεση λυθεί υπόψη. Θέλουμε αξιοπρεπείς ε, εργασιακές συνθήκες ε, και αμοιβή και αναγνώριση για τους οικιακούς βοηθούς και τους παρέχοντες φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οικιακή εργασία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη σύμβαση εργασίας και καθυστερημένες αμοιβέ, τις ατέρμονες ώρες εργασίας, χωρίς δικαιωμάτων αδειών, αρωτικών αδειών, κοινωνικών επιδομάτων ή αδειών άνευ αποδοχών. Είναι ιδιαίτερα επισφαλής αυτές οι θέση απασχόλησης ε, εξαιτία τη αποδυνάμωσης του κλάδου και τη επίθεση ε, κατά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επίση έχουμε αύξηση της ε, φτώχειας που καλύπτει στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή 30% του πληθυσμού εξαιτία των μακροοικονομικών πολιτικών και των πολιτικών λιτότητα που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ω απάντηση στην οικονομική κρίση. Οι πολιτικέ αυτέ προώθησαν την ιδιωτικοποίηση και την καταστροφή των κοινοφελών υπηρεσιών ε, και τη, της σε ηλικιωμένους παιδιά και ασθενείς. Και έτσι οι γυναίκες αναγκάζονται να παραμένουν στο σπίτι για να προσφέρουν αυτές τις φροντίδες. Αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδήγησαν σε εκμετάλλευση και φτώχεια και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τις επιβάλλει στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κυρία Γκονσάλες Πένιας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντρόφισσα Κωνσταντίν Κακούνερα για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε και για τη σωστή συνεργασία που είχαμε όλοι μαζί της στο εσωτερικό της Επιτροπής Απασχόλησης. Οι, οι απασχολούμενες οικιακές βοηθοί είναι οι γυναίκες που προστατεύονται λιγότερο από οποιασδήποτε άλλες εργαζόμενες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπάρξει σύμφωνα με την απόφαση 189 της ΔΟΕ πρόταση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αυτών γυναικών. Εργάζονται χωρίς καμία προστασία, έχουν τεράστια ωράρια, πολύ χαμηλές αμοιβέ, καμία εγγύηση για ασφάλεια και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Εμείς ζητάμε να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα αναγνωρίσει τη σημαντική αυτή απασχόληση έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή διαδικασία ενημέρωσης και επαγγελματικοποίησης της δραστηριότητας αυτής σε ένα πολύ μεγάλο προσωστό. Πρόκειται για γυναίκες, δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον για να αλλάξουν οι συνθήκες έτσι ώστε να καταστεί μια πιο συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόληση και να αναγνωριστεί ο ρόλος των οικιακών βοηθών στην κοινωνία μας. Το η Επίτροπος η κυρία Γιώροβα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Κούνεβα για την έκθεσή της που πραγματικά μας διαφωτίζει ε, για ένα τομέα που απασχολεί στον κόσμο 53 εκατομμύρια και στον κόσμο και 2,5 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση ε, τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Όπως λέτε πολύ σωστά ε, στην έκθεση, το 83% όλων των οικιακών βοηθών είναι γυναίκες. Είναι ένας γυναικοκρατούμενος αυτός ο τομέας και ε, Εστερνίζομαι πολλές από τις απόψεις και τις ανησυχίες σας. Για παράδειγμα, ανάγκη της αναγνώρισης του επαγγέλματος των οικιακών βοηθών και των παρεχόντων φροντίδα. Προκειμένου να μειώσουμε την αδήλωτη εργασία στον τομέα, να προωθήσουμε την ένταξή του στην αγορά εργασίας και να έχουμε μια αφύπνιση των κρατών μελών για το πρόβλημα και την ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών. Και μια και επιταχύνεται η γύραση του πληθυσμού, η ζήτηση για οικιακές εργασίες και παροχή φροντίδας πρόκειται να αυξηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει μια νέα αρχή για τους εργαζόμενους αγωνίες και τους παρέχοντες φροντίδα, γιατί στόχος μας είναι να λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις και τις οικογενειακές ανάγκες, τις ανάγκες των οικογενειών που έχουν εξαρτημένα άτομα, ηλικιωμένους και όχι μόνο τους γονείς, και να κάνουμε μια πιο δίκη χρήση των ε, ρυθμίσεων για τις ε, άδειες μητρότητας και πατρότητας. Είναι σημαντική και η ανάγκη επαγγελματοποίησης ε, του έργου των οικιακών βοηθών και παρεχόντων φροντίδα. Γι' αυτό θα προτείνουμε τρία σχέδια για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του κλάδου, την ποιότητα των υπηρεσιών και την παραγωγικότητα. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πλαίσιο που ξεκίνησε το 2012 για τέτοιε υπηρεσίες με στόχο να, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων που χρήζουν βοήθειας και φροντίδας. Επίσης, σημειώνω την ε, ε, αίτησή σας να αναλυθεί περισσότερο το θέμα της προστιθέμενης αξίας της πιθανής επαγγελματοποίησης ε, του κλάδου αυτού των οικιακών εργασιών. Η επαγγελματοποίηση των οικιακών βοηθών και των παρεχόντων φροντίδα στα νοικοκυριά θα αυξήσει την ελκυστικότητα του κλάδου αυτού και θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και επίσης θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Ε, μάλιστα το έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπηρεσιών που δίνονται κατοίκων και που δημοσιεύθηκε το 2012 αναγνωρίζει το δυναμικό σε θέση απασχόληση που έχει ο κλάδο αυτό, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τι οικιακέ εργασίε που παρέχονται στα νοικοκυριά και μάλιστα με χαμηλό κόστος ε, για τον δημόσιο κορβανά. Και από αυτή την άποψη τέτοιες διατάξεις που θα μεταφέρουν το κλάδο στην ε, νόμιμη οικονομία από την παραοικονομία θα πρέπει να ενθαρρυνθούν. Επίσης, σε ό,τι αφορά την πολιτική, ε, ε, η Γαλλία η και το Βέλγιο έχουν αντιστοιχείς διατάξεις, αντίστοιχα σερβίς και η Σουηδία έχει προβλέπει κάποιες φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις για να προωθήσει τέτοιες ε, υπηρεσίες. Επίσης, ε, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι σημαντική προτεραιότητα για τους οικιακούς βοηθούς και τον τους παράγοντες φροντίδας, γιατί όλοι θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις δεξιότητες. Αυτό θα βελτιώσει και την, τις πιθανότητες ε, ανέβρες εργασίας και γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη βελτίωση της διαφάνειας των προσόντων και των δεξιοτήτων. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και για τους μετανάστες αλλά και για τους πρόσφυγες προκειμένου να ενταχθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας. Σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τη Σύμβαση για την δίκαιη και αξιοπρεπή εργασία για τους οικιακούς βοηθούς, τη Σύμβαση Περιθμών 189, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ συχνά ε, προώθησε την κύρωση και το Σεπτέμβριο του 2015 με τη Λουξεμβουριανή Προεδρία καλέσαμε τα κράτη-μέλη να κυρώσουν την Σύμβαση 189 της ΔΟΕ. Και συμμεριζόμαστε την έκκλησή σας για ένα κατάλληλο επίπεδο υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό χώρο για τους εργαζόμενους στο κλάδο των οικιακών εργασιών. Γιατί ο αποκλεισμό των οικιακών βοηθών από το πεδίο εφαρμογή οδηγία 89-391 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την υγεία και προστασία των εργαζομένων θα εξεταστεί μετά την αξιολόγηση του κοινοτικού κεκτημένου υπό το πρίσμα της υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Όπως αναφέρετε και εσείς στην έκθεσή σας, πρόσφατα τα τελευταία χρόνια είχαμε αύξηση του ποσοστού των μεταναστριών ε, οικιακών βοηθών. Και σημειώνουμε τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν νόμιμα εισοδήματα για τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίσουν στοχευμένα μεταναστευτικά προγράμματα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ένα, ε, ξεκινήσει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα ένταξης για τους μετανάστες εργαζομένους που περιλαμβάνει και πιλωτικά προγράμματα προκειμένου να βοηθηθούν οι μετανάστες και οι βοηθοί στην Ευρώπη. Σημερίζομαι και τις ανησυχίες σας για την αδήλωτη εργασία τα επίπεδα της είναι υψηλά στο κλάδο αυτό και επηρεάζει αρνητικά τις εργασιακές συνθήκες των ανθρώπων αυτών, την ποιότητα των υπηρεσιών τους και γενικότερα επηρεάζει αρνητικά και την οικονομία. Η επισημοποίηση λοιπόν, η επαγγελματοποίηση των εργασιών αυτών θα εξασφαλίσει κοινωνική προστασία και θα αυξήσει ε, και το εισόδημα του κράτους. Επίσης θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που συνδέεται αναπόσπαστα με τις εργασιακές συνθήκες και την αναγνώριση των προσόντων τους και δεξιοτήτων τους. Πιστεύω ότι η νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη διεύρυνση της συνεργασίας, για την πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας θα συμβάλλει στην αφύπνιση, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και ανάλυση των εμπειριών προκειμένου να βρεθούν οι λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και χαίρομαι που επισημαίνεται το σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις ε, στο τομέα των οικιακών εργασιών και παρόχης φροντίδας. Θα πρέπει φυσικά να ε, γίνει σεβαστή και η αυτονομία. Ε, θα πρέπει να υπενθυμίσω την πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να στρέψει την Ευρώπη προς μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Κανένας δεν θα πρέπει να μείνει πίσω περιθωριοποιημένος και αυτή η έκκληση περιλαμβάνει και τους οικιακούς βοηθούς. Είναι πολύ επίκαιρη λοιπόν η έκθεσή σας και θα μας βοηθήσει να προδεύσουμε σε πολλές πολιτικές και να τις συνδυάσουμε μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ. Κλείνει η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο.